Allora io comincio con questo, vero Maria? Con questo e poi vi passo io l'approvazione del processo verbale. Sì. Possiamo cominciare. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας πρέπει πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, επί της οποίας σας ανακοινώνω ότι τα σημεία 9 και 33 ε, δεν θα μας απασχολήσουν. Προτείνω να ξεκινήσουμε ε, με μία επιστολή η οποία αφορά την ε, δημόσια πρόσβαση των, ε, ε, του κοινού στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αργότερα να το κάνουμε, εντάξει, της κυρίας Λίχτεμπεργκ. Σας λέγω επίσης ότι λόγω τεχνικών ε, προβλημάτων στο Eurostar η κυρία Γιώ Wallis ε, θα φτάσει με ε, ελαφρά καθυστέρηση και επομένως τα σημεία 5 και 6 θα μας απασχολήσουν αργότερα όταν δηλαδή θα έρθει η κυρία Wallis. Με αυτές τις τροποποιήσεις εγκρίνεται η μέρη σε διάταξη, πάρα πολύ ωραία. Περνούμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών ε, της συνεδριάσεως της 20 και 21ης Ιουνίου 2011 καθώς επίσης ε, και της 11ης και 12ης Ιουλίου 2011. Παρατηρήσεις επί των πρακτικών όχι, επομένως θεωρούνται εγκεκριμένα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, είναι το σημείο 4, δηλαδή έκθεση η οποία αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 89 κάθετος 666, 2005-56 και 2009 κάθετος 101 ε, όσον αφορά τη διασύνδεση των εμπορικών, κεντρικών και λοιπόν μητρών των επιχειρήσεων. Η συγητής είναι ο κύριος Λέχνας, τον οποίο δίνω και τον λόγο αμέσως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα στην διαβούλευση για το πράσινο βιβλίο μιλήσαμε ήδη για το θέμα αυτό είχαμε εγκρίνει και ψήφισμα και μετά από την κατάθεση της προτάσεως συζητήσαμε σύντομα. Εδώ μεταξύ μας δεν υπάρχει α, καμία αμφιβολία ότι η διασύνδεση αυτή είναι σημαντική και ορθή και πρέπει να προχωρήσει. Σημειώνονται δύο τομείς προβλημάτων. Αφενός επί της ουσίας και το άλλο, και το θέμα αυτό είναι σημαντικό, είναι το τεχνικό θέμα. Εγώ είπα ότι προσωπικά δεν έχω τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την χρήση αυτών των πλατφορμών και για το ποια ψηφιακά και άλλα προβλήματα σημειώνονται. Και νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο, όχι ως συνάδελφοι, αλλά ως θεσμικό όργανο, δεν διαθέτει και αυτό εμπειρογνωμοσύνη. Επίσης, θεώρησα ότι ήταν σωστό να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε την αρχή για να δούμε αυτό το βλέποντας και αποφασίζοντας. Να δούμε δηλαδή πού πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χαρακτήρα τεχνικού ή πρακτικού. Η Πολωνική Προεδρία στο μεταξύ, στον φάκελο αυτό, έχει δράσει με πολλή αποφασιστικότητα και έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις και στο Συμβούλιο, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει στην σύνταξη ενός κειμένου, το οποίο μου διαβίβασαν, το εξήτασα και είδα σε ό,τι αφορά το ψήφισμά μας αλλά και την προσωπική μου γνώμη ότι επί της ουσίας έχει οριμάσει πλέον η απόφαση και μπορεί να προχωρήσει αλλά ορισμένα τεχνικά βρίσκονται ακόμα σε διαδικαστική φάση και δεν μιλώ για τη διαδικασία της νομοθεσίας αλλά του τελικού καθορισμού. Και για να προχωρήσουμε έχω συντάξει την έκθεση αυτή σε αγγλική γλώσσα Είναι όμως περιορισμένη η γνώση μου της αγγλικής γνωρίζω όμως την τεχνική ορολογία μπορώ να την κατανοήσω και να την επαληθεύσω. παρέμεινα στα πλαίσια των εγγράφων της Πολωνικής Προεδρίας και έρχομαι στα τεχνικά θέματα. Είναι σαφές, όπως άλλωστε τα είχαμε εγκρίνει και στη συζήτηση του Πράσινου Βιβλίου, ότι μπορεί να γίνει μια πλατφόρμα για μια πύλη πρόσβασης και όχι νέο, νέα ευρωπαϊκή καταχώρηση. Θα πρέπει το φορμά να είναι στάνταρτ επειδή το θέμα των γλωσσών είναι σημαντικό, δεν γνωρίζω ακριβώ πώς μεταφράζεται ούτε και στα γερμανικά, ενώ ότι το index που θα πρέπει να είναι αυτή η επικεφαλίδα, το αρχικό τμήμα, σε όλες τις γλώσσες, ώστε ο ενδεχόμενος χρήστης να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και να παραμείνει μέσα στα πλαίσια των εθνικών γλωσσών. Το δε σύστημα να υπαχθεί ολόκληρο την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μην φύγει δηλαδή εντελώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτά τα μητρώα είναι πολύ σημαντικά και από, τη, από αυτά εξαρτώνται πολλές και σημαντικές νομικές αποφάσεις. Αυτό βέβαια είναι εξασφαλισμένο τώρα. Επομένως, την ευθύνη αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μπορεί η ίδια να αποφασίσει κατά πόσον θα αναθέσει περαιτέρω το έργο αυτό, ενδεχομένως σε ιδιωτικούς φορείς. Αλλά την ευθύνη εξακολουθεί να την φέρει η ίδια καθώς και για το σύστημα αναζήτησης. Σημαντικό επίσης είναι οι διάφορες νομικές έννοιες αναλόγως με τα διάφορα εμπορικά μητρώα, τα εθνικά εμπορικά μητρώα δηλαδή, περιλαμβάνεται, να περιλαμβάνεται ότι δεν θα πρόκειται να χρειαστεί έξτρα γραφειοκρατική προσπάθεια. Τώρα, το χρηματοδοτικό έχει περιοριστεί. Έχει είχαν προβλεφθεί προθεσμίε των 15 ημερών που μου φάνηκε εμένα ότι δεν ήταν ορθό και γι' αυτό έβαλα τη λέξη αμελητή ώστε να είναι σαφές τώρα το πόσο κωδικός θα διαμορφώνεται αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο έγγραφο η Κομισιόν όπως και σε πολλές άλλες νομοθετικές πράξεις που υποβάλλει τελευταία έχει βάλει πολλές κατεξουσιοδότηση και εγώ το επέκρινα αυτό και στην ε, ΙΜΚΟ. Βέβαια υπάρχει τώρα μια δυσκολία, την οποία τονίζω ρητά. Εγώ προσπάθησα από την πλευρά μου και παρακάλεσα και την Πολωνική Προεδρία να κάνει σχετικές ενέργειες να μπουν στο νομοθετικό κείμενο όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Βέβαια δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δηλαδή ε, δυνατόν, δυνατόν να καταγραφούν τα πάντα εκεί, διότι πολλά θα προκύψουν από τη χρήση στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Δεύτερο, ίσως θα εκπλήξει αυτό ορισμένους, πρότεινα από την πλευρά μου και δέχομαι άλλωστε ένα μέρος να επιλύεται μέσω πράξεων κατά αλλά και ένα άλλο με εκτελεστικές. Ίσως αυτό να μην είναι σαφές για όλους. Στις πράξεις κατά αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν της δικής της διεξουσίας. Εγώ έχω προβλέψει τώρα τρεις μήνες, οι δύο μήνες ήταν πολύ περιορισμένοι, έχει τη δυνατότητα της ανάκλησης. Αλλά ποιο θα το κάνει αυτό. Με τι εκατοντάδε τέτοια κείμενα το κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Τώρα όμω για τι εκτελεστικέ πράξει είναι διαφορετικά. Όπω προβλέπετε τώρα, καλούνται να συμφωνήσουν οι χώρε μέλη. Και επειδή τα πράγματα εδώ είναι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα, και μόνο σε συνεργασία με τι χώρε μέλη, με τα δικά του μητρώα και με τι δικέ του τεχνικέ προδιαγραφέ είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται να δείξουμε και κάποια εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν η Κομισιόν και η χώρα μέλο η ίδια είναι πεπισμένε ότι στα πλαίσια τη εκτελέσεω είναι ενδεδειγμένη μια συγκεκριμένη τεχνική διαδικασία, αυτό να γίνεται δεκτό. Εδώ, εν προκειμένου, το Κοινοβούλιο δεν θα έχει την δυνατότητα αυτό βέβαια το γνωρίζω, αλλά εκ του αποτελέσματος και επί της ουσίας βρίσκω ότι αυτό είναι ενδεδειγμένο και επιβεβλημένο, γιατί πρόκειται για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, όπου το Κοινοβούλιο εν τέλει δεν μπορεί παρά να συγκατανεύσει. Και για μένα αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι οι χώρε μέλη με του δικού του εμπειρογνώμονε και που γνωρίζουν τα δικά του προβλήματα να συμφωνούν και εκεί να αρκούμεθα. Σε αυτό αυτόν αρκούμεθα δηλαδή. Ο βασικός λόγος, από ό,τι κατανοώ και που δεν είναι το κείμενο απόλυτα ίδιο με αυτό που συζητήθηκε στο Συμβούλιο, εγώ σε ορισμένε περιπτώσει, έβαλα και τη δική μου προσωπική σκοπιά, παρόλα αυτά σε μεγάλο βαθμό ήδη έχει συνενέσει η πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Αναμένουμε τώρα τις μεταφράσει και μετά θα ξανασυζητήσουμε εκτενώς επί της ουσίας. Εγώ βέβαια επιφυλάσσομαι να προχωρήσει τη συζήτηση αυτή. Ο στόχος μου ήταν τώρα, αφού και η Πολωνική Προεδρία έχει καταβάλει τόσες προσπάθειες, να δοθεί η δυνατότητα να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Λέχνερ. Μου φαίνονται πάρα πολύ σωστές ε, οι παρατηρήσεις σας. Θα ξεκινήσει λοιπόν ανταλλαγή απόψεων. Η Εύελιν Μπρέχνερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, πολύ σαφή παρουσίαση κύριε Λέχνερ. Ορισμένες συμπληρώσεις. Βέβαια, καλούμαστε εμείς εδώ, τώρα όσοι δεν έχουμε αυτή την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, και σε ένα θέμα επάνω το οποίο είναι τόσο σημαντικό γιατί έχει πολύ σημαντικές πρακτικές επιπτώσεις τόσοι συμβολογράφοι, δικηγόροι και ούτω καθεξής θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτές. Άρα, ζητείτε να δείξουμε τώρα εμπιστοσύνη. Θα έλθω σε ορισμένα από τα σχόλιά σας. Πρώτα για την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των χωρών μελών που αναφέρατε. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι κέριο αίτημα. Όταν προχωρούμε σε μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι χώρες. Και ορισμένα άλλα που είπατε. Αυτή η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη την οποία δεν διαθέτουμε και είναι δικαιολογημένη. Να φύγουν δηλαδή οι delegated acts από εδώ και να έχουμε πιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως και στις χώρες μέλη, ότι στην εκτέλεση θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Εγώ ευχαρίστω θα ήθελα να υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη και ιδίω απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία βρίσκονται και οι εμπειρογνώμενε. Ωστόσο, ως βουλευτής δεν θέλω να πω ότι είμαι καταρχήν δυσπιστή, αλλά είμαι κάποιο επιφυλακτική σχετικά με αυτά και ιδίω όταν δεν λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι η ίδια εκείνη η οποία θα χειρίζεται το δίκτυο αυτό, αλλά αυτό ανατίθεται σε τρίτους. Αυτός ο συνδυασμός με καθιστά επιφυλακτική. Διότι θέματα όπως αυτό απαιτείται να έχουν έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Για την τροπολογία σας είπα 21 όπου ζητείτε εσείς τη διαγραφή στην παραπομπή στην προστασία των δεδομένων. Αυτό έχει σχέση με την επερχόμενη νομοθεσία διακόπτη μετά από νεύμα του κ. Λέχνερ. Καλά, θα το συζητήσουμε λοιπόν, ναι, μεταξύ μας. Όπως είπαμε λοιπόν, η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των χωρών μελών. Θέλω να το τονίσουμε ιδιαίτερα αυτό στο τέλος, εφόσον θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι από τα κέρια αιτήματα. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ, Εύελιν. Άλλη... Άλλες παρεμβάσεις, όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπω θέλει να σχολιάσει, θέλει να πει κάτι. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Επομένω, ολοκληρώσαμε την εξέταση αυτού του σημείου. Περνούμε στο επόμενο σημείο. όπω είπαμε και προηγουμένω, τα σημεία 5 και 6 της ημερησία διατάξεω ε, θα μα απασχολήσουν λίγο αργότερα, ε, διότι η κυρία Wallace δεν έχει φτάσει ακόμα. Σημείο 7, λοιπόν, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το εξή θέμα, αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας ε, σε, των πολιτών. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο να μου πει εάν μπορεί να μιλήσει από κοινού για τα σημεία 7 και 8 γιατί είναι ε, εισηγητής και για το σημείο 8 το οποίο αφορά τα ελάχιστα, την ελάχιστη κοινή συνεννόηση για τα δικαιώματα, τη στήριξη, την προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Ναι, συμφωνώ κύριε Πρόεδρε, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το σημείο 7, τον κανονισμό δηλαδή, που εντάσσεται στο πακέτο για την προστασία των θυμάτων που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου τρέχοντος έτους, που περιλαμβάνει δύο ε, μηχανισμούς, ε, δύο νομοθετικές πράξεις, τον κανονισμό για τον οποίο είμαι εισηγητής επί της ουσίας και μια οδηγία για την οποία είμαι συντάκτης γνωμοδότησης και αφορά το σημείο 8 της ημερήσης διάταξης. Ο κανονισμός για τον οποίο θα εκπονήσω έκθεση συμπληρώνει ουσιαστικά την ΕΠΟ, την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, που ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 2009 σε πολλές χώρες και κανονικά θα εφαρμοζόταν σε ποινικά θέματα. Πρόκειται για ένα νέο μέσο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρατείνει την αναγνώριση των μέσων προστασίας των θυμάτων και στις αστικές υποθέσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ την άποψη αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση του σχετικού μέτρου, που αναμφίβολα θα συμπληρώσει την προστασία στα θύματα, Φέροντα τα θύματα στο επίκεντρο των πολιτικών και των ε, ανησυχιών και της μέρημνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά τη γνώμη μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναμειχθεί ενεργά στη διαδικασία αυτή. Θέλουμε να συμπληρώσουμε την πρωτοβουλία των 100 μελών του Σεπτεμβρίου του 2009 της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας και τη συμπληρώνει με ένα νέο μέσο ε, αμοιβαίας αναγνώρισης ε, προληπτικών ε, μέτρων και μέτρων προστασίας για προστασία ενός θύματος όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την σωματική ψυχική του ακυρεότητα ή τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία το μεταμηχανισμό αυτό και με βάση την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών και εξώδικων πράξεων προβλέπεται αυτόματη και εύκολη αναγνώριση που εξασφαλίζει τα μέτρα προστασίας που έχει αποφασίσει ο Εθνικός Δικαστής χωρίς να μεσολαβούν άλλοι. Γίνεται αυτόματη αναγνώριση και νομίζω ότι έτσι εξοικονούμε και χρήματα και χρόνο με την διαδικασία, γιατί δεν χρειάζεται πια η διαδικασία εξεκουάτορ της έκδοσης εκτελεστήριου τίτλου. Σίγουρα θα γίνουν πολλές συζητήσεις ε, για τα πιστοποιητικά για παράδειγμα και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα πιστοποιητικά, αλλά νομίζω ότι είναι ε, καλή ευκαιρία αυτή για να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων και τα σχόλιά τους για το θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κανονισμό, σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα να πω ότι είμαι ανοιχτός και διαλλακτικός. Περιμένω τις προτάσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Κατά πάσα πιθανότητα θα καταθέσω το σχέδιο έκθεσή μου πριν τα Χριστούγεννα, ώστε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στα τέλη Μαρτίου και στην Ολομέλεια του Απριλίου ή του Μαΐου. Κατά προτίμηση την Ολομέλεια του Απριλίου. Επαναλαμβάνω, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Τώρα το σημείο 8 οδηγία για την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Θα ήθελα να πω για την οδηγία αυτή ότι η οδηγία για την οποία θα κληθούμε να συντάξουμε γνωμοδότηση στην ε, Επιτροπή μας ε, με οριζόντιο τρόπο προβλέπει κάποια δικαιώματα υποστήριξη και προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων χωρί διακρίσει. Και επίση ε, κατοχυρώνει θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων με την πρόταση αυτή. Ε, δικαίωμα λήψης ενημέρωσης για την ε, περίπτωση αυτή. Από την πρώτη επαφή με τις αρμόδιες αρχές έχει δικαίωμα μετάφρασης, διερμηνίας, ε, να καταλαβαίνει και να γίνεται κατανοητός. Υποστήριξη των θυμάτων, δικαίωμα δωρεάν δικαστικής αρρωγής, επιστροφή εξόδων. Πολλά και διάφορα δικαιώματα που αναπαριθμούνται στην οδηγία αυτή και δεν προλαβαίνω τώρα να σας τα αναφέρω. Πολύ σημαντική είναι η εισαγωγή τις έννοιες του σεβασμού του θύματος, ώστε να μην γίνει περαιτέρω θυματοποίηση αυτών των ανθρώπων. Επίσης, ε, βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και το θέμα της αποζημίωσης και της αποκατάστασης είναι πολύ σημαντικό. Συμπεριλαμβάνονται πολύ σημαντικά σημεία για την βοήθεια και υποστήριξη των θυμάτων, τόσο και από ποινική άποψη, όσο και από οικονομική, ψυχολογική και ιατρική αρρωγή. Και νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή και καλό θα ήταν να την συζητήσουμε κι εμείς. Μία παρατήρηση έχω μόνο και θα ήθελα να πω με κάποια θλίψη γιατί είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μου. Εκφράζω τη θλίψη μου γιατί ε, παραμερίστηκαν κατά κάποιο τρόπο τα θύματα της τρομοκρατίας. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάτι 8 Μαΐου που συνοδεύει αυτό το πακέτο προς μέτρων για την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων, στο σημείο 4 για τι ειδικέ κατηγορίε θυμάτων, περιλάμβανε και τα θύματα τη τρομοκρατία στην ομάδα προστασία. Παρ' όλα αυτά, τα θύματα της τρομοκρατίας ε, αναφέρονται και στο τμήμα 3 του άρθρου 18, αλλά στη συνέχεια, στο άρθρο 18, που μιλά για την ταυτοποίηση των ευάλωτων θυμάτων ε, παραμερίζονται, αγνοούνται. Πολύ σωστά στο σημείο εκείνο αναφέρονται τα ενηλικά άτομα, τα άτομα με αναπηρίες, τα θύματα σεξουαλικής βίας, τα θύματα εμπορίας α, ανθρώπινων όντων. Είναι σίγουρα ευάλωτα αυτά τα βήματα, αλλά γιατί παραλείπονται τα θύματα της τρομοκρατίας από τα ιδιαίτερα ευάλωτα αυτά θύματα. Λυπούμε που προβαίνει σε αυτή την παράληψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να το επισημάνω για να γίνει σχετική συζήτηση και να δω αν συμφωνούν και οι συνάδελφοι με την πρωτοβουλία μου αυτή, να συμπεριλάβουμε και τα θύματα της τρομοκρατίας στο κατάλογο με τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα. Ίδιο χρονοδιάγραμμα με αυτό του κανονισμού προβλέπεται για την γνωμοδότηση. Θα την υποβάλω πριν τα Χριστούγεννα, ώστε το συντομότερο δυνατό να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Επαναλαμβάνω, είμαι ανοιχτό και περιμένω τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας. Φυσικά περιμένω και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που από ό,τι ξέρω ε, είναι παρούσα εδώ στη συνεδρίαση. Θα ήθελα να συνεργαστούμε στενά ώστε και η έκθεση και η γνωμοδότησή μας ε, να έχουν ε, βάρος, να είναι σημαντικές και χαίρομαι που και τα δύο θέματα βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση των δύο εκθέσεων. Επιθυμεί κάποιος να πάρει το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως. Ναι, όχι. Όχι. Ωραία. Εντάξει, ολοκληρώνουμε λοιπόν και την εξέταση αυτού του σημείου και περνούμε στο επόμενο που αφορά πάλι την κυρία Νταϊάννα Wallis, η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα, άρα περνάμε στο 10 της Εύλιν Ρέγνερ. 14η οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά έδρας ε, των επιχειρήσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προχωρείτε γρήγορα κύριε Πρόεδρε. Στη νομική επιτροπό, επιτροπή το θέμα της μετεγκατάστασης δεν είναι και κανένα καινούριο θέμα. Μέχρι τώρα έχουμε πει ότι μια σχετική οδηγία θα πρέπει να γίνει το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην προηγούμενη θητεία της Ευρωβουλής. Ψηφίστηκε δηλαδή τον Ιανουάριο του 2009 η έκθεση του κυρίου Λένε. Άρα έχουμε μια βάση. Ορισμένα πράγματα έχουν αλλάξει. Στην Ευρώπη της ενιαίας αγοράς στην περίπτωση μετεγκαταστάσεως των επιχειρήσεων θα πρέπει βεβαίως να διαλύσουν τα πάντα οι ε, επιχειρήσεις και να ξαναστήσουν την επιχείρησή τους αλλού. Αυτό βέβαια έχει υψηλό ε, κοινωνικό κόστος, έχει συνεπάγεται γραφειοκρατικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Πράγματα δηλαδή που καθιστούν απαραίτητη την έκδοση σχετικής οδηγία. Και αυτό είναι και το κύριο μήνυμα της εκθέσεώς μου, δηλαδή η προτροπή στην Ευρωπαϊκή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί νομοθετικά. Ορισμένα από τώρα από τα θέματα που θίγω είναι τα εξή. Θέτω ευθέως το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Το θέμα της έδρας. υπάρχει μέγα πρόβλημα αξιοπιστίας της Ευρώπης. Δηλαδή και οι επενδυτές αλλά και οι φορολογούμενοι όταν θέλουν να επενδύσουν σε διάφορα hedge fund ή αλλού θέλουν να γνωρίζουν τι είδους επιχείρηση είναι αυτή. Υπάρχουν επιχειρήσεις που με δική τους διεύθυνση είναι ένα ταχυδρομικό κουτί. Τα πράγματα λοιπόν πρέπει να λεχθούν με το όνομά τους. όπως δεν είχε πράξει ο τότε Επίτροπος Μαγκρίβη. Δηλαδή πρέπει να διακριθεί η μετεγκατάσταση της πραγματικής έδρας από την διοικητική. Λοιπόν, σημειώνω βεβαίως και την υποχρέωση κοινοποίηση που περιλαμβόταν και στην έκθεση Ελένε, καθώς και το δικαίωμα συναπόφασης των εργαζομένων, όπου ήδη υπάρχει μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχολήσεως και γι' αυτό και την αναφέρω και στην παρούσα Επιτροπή. Εκεί λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση εγκρίθηκε με τεράστια πλειοψηφία, με μόνο μία ψήφο κατά. Για θέματα δηλαδή συναποφάσεως στη βάση των υφισταμένων ε, διατάξεων της ε, Ευρωπαϊκής Κεφαλαιοχικής Εταιρείας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι και εγώ. Θα αρκεστώ σε αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις για την εκθεσή μου. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, στις 20 Δεκάτου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 23 Ενδεκάτου. Το οποίο με ικανοποιεί γιατί γνωρίζω ότι θα υπάρξουν και Άλλε απόψει. Αναμένω λοιπόν μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και σύνταξη της εκθέσεως που ελπίζω εν τέλει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί νομοθετικά. Ευχαριστώ, Εβελίν. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μας έκανες. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Κανείς. Κανείς. Και εδώ εμείς στρεφόμαστε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως κανείς δεν θέλει. Δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα όλοι, είναι Δευτέρα. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 11. 11. Σεμπαστιάν Βαλεντίν Μπόντουι, εισηγητής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση των Εταιριών. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το δίκαιο αυτό στις ε, μεγάλες ε, εταιρείες και τις ε, εισηγμένες στα χρηματιστήρια. Ε, υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες ε, οι οποίες είναι σημαντικές ακριβώς ε, λόγω της μονοπωλιακής τους θέσης ή λόγω του τζίρου που έχουν. Όμως δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί το ζήτημα αυτό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται κάποια ελευθερία κίνησης. Θα εμπνευστώ στη, από την Πράσινη Βίβλο. Όσον αφορά λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορώ να πω το εξής. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εκτελεστικό ε, διευθυντή. Αυτές οι δύο θέσεις ε, θα πρέπει να είναι διαφορετικές και να καλύπτονται από διαφορετικούς ανθρώπους. και εμείς ε, δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου ε, με την εκτελεστική διεύθυνση. Όσον αφορά τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να απαρτίζεται από άτομα με ε, αποδεδειγμένη εμπειρία στα θέματα και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν δεν θα υπάρχει ε, πρόβλημα όσον αφορά τις ε, άλλες τους δραστηριότητες και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να συμμετέχουν και στην εκτελεστική διοίκηση επίσης να παρακολουθούνται ε, ότι δηλαδή συμμετέχουν σταθερά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι δεν συμμετέχουν απλώς μια φορά και μετά κάθονται στο σπίτι τους. Το θέμα της ε, διαφοροποίησης είναι πολύ σημαντικό, καθώς επίσης ε, και το θέμα των μη μονίμων κατοίκων. Σημαντικό και αυτό και των μη υπηκών. Επίσης, ε, ο αριθμός των γυναικών θα πρέπει να αυξηθεί, χωρίς όμως να πιστεύω ότι θα πρέπει να καθοριστούν υποχρεωτικές δεσμευτικές ποσοστώσεις διότι στην ουσία οι ίδιοι οι μέτοχοι αποφασίζουν και επιλέγουν ε, αυτούς που θέλουν να ε, ε, επιλέξουν στα διοικητικά συμβούλια. Να γίνουν λοιπόν κάποιες προτάσεις, όχι υποχρεωτικές, αλλά ευέλικτες. Επίσης, η ίδια η εταιρεία να μπορεί ε, να δώσει, να κάνει κάποιες προτάσεις ε, για τον αριθμό γυναικών ε, που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να πει δηλαδή μέχρι ποιο μέγιστο αριθμό γυναικών μπορεί να φτάσει. Δηλαδή Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις ε, στις οποίες δεν μπορεί να επιβληθεί ας πούμε ένα ποσοστό 40%. Εκεί ε, μπορεί να δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα και επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν αρχικά τουλάχιστον να δοθούν κάποιοι ευέλικτοι στόχοι και να πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει τον στόχο όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών. Για τους διαχειριστές τώρα Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και αυστηρούς κανόνες αλλά και έναν κώδικα συμπεριφοράς όσον αφορά τον αριθμό των θητιών που μπορεί κανείς να συσσωρεύσει ε, και που να μην μπορεί ας πούμε να ξεπεράσει ε, τις πέντε θητείες. Αυτό το λέω τώρα σαν παράδειγμα. Να μην μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να, είναι, να ασκήσει πάνω από πέντε θητείες και για αυτούς που προτίθενται να ε, υπερβούν ε, τις πέντε θητείες, ε, τότε θα πρέπει να εξηγηθεί σε όλους τους μετόχους δημόσια οι λόγοι για τους οποίους επελέγει ξανά ο ίδιος επικεφαλής. Έτσι ώστε και το, και το κοινό αλλά και οι κυβερνήσεις και τα συμβούλια να καταλαβούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται ξανά το ίδιο άτομο. Ε, άλλα προβλήματα δεν βλέπω να υπάρχουν. Πάντως, και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τον εκτελεστικό διευθυντή θα πρέπει να αποφασίζει η Ολομέλεια των Μετόχων. Όμως δεν συμφωνώ ε, με τον καθορισμό ανωτά του ορίου αμοιβών. Ε, η ίδια η Γενική Συνέλευση των Μετοχών θα πρέπει να πάρουν την απόφαση. Ε, θα πρέπει στην ουσία όμως να πάρει απόφαση για, τον, την μεθοδολογία, για την μέθοδο μάλλον υπολογισμού της αμοιβή των στελεχών και όχι αποφάσεις για συγκεκριμένα ε, αριθμητικά στοιχεία γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε και την ιδιωτική ζωή αυτών των ανθρώπων. Επίσης, ε, ε, πιστεύω ότι το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει και στις διαδικασίες αυτές. Θα πρέπει επομένως να ενισχυθεί ο, ο ρόλος ε, και των διαφόρων επιτροπών, είτε πρόκειται επιτροπή ε, μισθοδοσίας, είτε πρόκειται για, για τον οικονομικό έλεγχο, επιτροπή οικονομικού ελέγχου κτλ. Και αυτές οι επιτροπές θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος των μετόχων βεβαίως είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι. Όμως ε, πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει ε, να ενισχυθεί και ο ρόλος των διαχειριστών το λέω αυτό με την έννοια ότι βεβαίως είναι σημαντικός ο ρόλος των μετόχων, αλλά μπορεί οι μέτοχοι να μην θέλουν ε, να συμμετέχουν περαιτέρω στις διαδικασίες. Έχουμε επίσης διάφορες, διάφορα στοιχεία όπως είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ε, για ορισμένες ε, ε, εταιρείες. Δεν συμφωνώ όμως με, τον, με την υποχρεωτική ψήφο γιατί οι ίδιοι οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν, θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν ναι ή όχι θέλουν να ψηφίσουν. Οι μέτοχοι θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους ενώ υπάρχουν χώρες στις οποίες απαγορεύονται οι συμφωνίες μεταξύ των μετόχων. Αντιθέτως εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως θεμητό και νόμιμο να συνεργάζονται και να συνεννοούνται οι μέτοχοι μεταξύ τους πριν φτάσουν στη Γενική Συνέλευση. Όσον αφορά τώρα ε, ε Όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, ε, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει οι κανόνες που θα εφαρμοστούν να είναι αυστηροί. Όταν έχουμε λοιπόν συναλλαγές μεταξύ μερών που έχουν ίδια ε, συμφέροντα, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ανακοινώσουν ε, ότι ακριβώς υπάρχει αυτή η σύγκρουση συμφερόντων και επομένως να ακυρωθούν οι ε, συναλλαγές. Επίσης, οι μικροί μέτοχοι θα πρέπει να μπορούν να αντιδράσουν σε περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων τους από τους μεγαλομετωχούς μετόχους. Επίσης να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρξει κατάχρηση εξουσίας. Όσον αφορά τώρα τους συμβούλους, ε, και την, ε, αυτά τα συμβόλαια stewardship ε, πρόκειται για συγκεκριμένες συμβάσεις με εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τις ψήφους των μετόχων πιστεύω ότι η δυνατότητα συλλογής των μη εκπεφρασμένων ε, ψήφων θα πρέπει οι εταιρείε αυτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικές ε, και στην προκείμενη περίπτωση επίσης θα πρέπει να δούμε εάν ε, ε, έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων γιατί αυτές οι εταιρείε οι οποίες συλλέγουν τις μη εκποφρασμένες ψήφους θα πρέπει να προσέχουν και να ανακοινώνουν τις περιπτώσεις συγκρούσεων ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων. Επίσης, πιστεύω ότι εδώ δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικές αρχές ε, γιατί είναι πιο εύκολο όταν υπάρχουν ευέλικτοι κανόνες οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν. Είναι καλύτερα να προσπαθούμε πάντα ε, να έχουμε εξηγήσει από τους μετόχους και όχι να τους επιβάλλουμε υποχρεώσεις. Οι κανόνες επίσης ε, ε, και τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σαφή. Σε περίπτωση δε μη τήρησης του κανόνος θα πρέπει η εταιρεία να εξηγήσει σαφώς γιατί απομακρύνθηκε από αυτόν τον κανόνα. Τέλος, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ανάλυση λειτουργίας ε, της ε, εταιρείας από, μια, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ε, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι εταιρείες αλλά να μην είναι υποχρεωμένες να προστρέξουν σε αυτόν τον κατάλογο. Ε, και σε αυτόν τον έλεγχο αλλά βεβαίως να πούμε ότι ε, οι εταιρείες οι οποίες θα έχουν αυτό το πιστοποιητικό ε, θα έχουν την δυνατότητα να έλξουν περισσότερα κεφάλαια αλλά εν πάση περιπτώσει να αφήσουμε ελεύθερη την εταιρεία να αποφασίσει. Εγώ θα στείλω το έγγραφό μου και στους κοιόδης εισηγητές και θα καθορίσουμε και τις προθεσμίες. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Η Εύελιν Ρέγνερ έχει το λόγο. Ähm, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Ωστόσο, θέλω να πω κάτι ουσιώδες. Μιλούμε τώρα για corporate governments στα πλαίσια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και δεν μπορούμε βέβαια να μείνουμε στα business as usual, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου λόγω οικονομικής κρίσεως βλέπουμε πράγματα που πραγματικά είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό και θέλω να υπενθυμίσω αυτή την βασική αρχή. Ό,τι βασίζεται στην οικειοθελή δράση δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν λειτουργεί ποτέ, αλλά συχνά δεν λειτουργεί σωστά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και να αναφερθούμε ιδιαίτερα σε όλα όσα δεν είναι μόνο εθελούσια αλλά και σε όσα μπορούν να ελέγχονται καθώς και να ε, επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις. Για παράδειγμα, Αυστρία αξιολογήθηκε η εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς με αποτέλεσμα στη μικρή μας χώρα όπου ορισμένες εισηγμένες επιχειρήσεις, τέσσερις, τέσσερις τήρησαν τους κανόνες και 263 όχι. Βλέπουμε λοιπόν την ανάγκη να δραστηριοποιηθούμε και πέραν από οποιουσδήποτε εθελοντικούς κανόνες να ισχύσουν άλλοι δεσμευτικοί. Και έρχομαι τώρα στις ποσοστώσεις Γνωρίζω ότι στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και να υποστηρίξουμε τις προτάσεις Reading, όπως για την Corporate Governance και όλες τις άλλες προτάσεις που οδηγούν σε περισσότερη διαφοροποίηση είτε με συμμετοχή εκπροσωπών, εκπροσώπων των εργαζομένων ή με όλους εκείνους οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούνται στις επιχειρήσεις και να μην είναι απλώς μια κλειστή λέσχη. Με την έννοια αυτή χαίρομαι από τώρα για τις ε, μελλοντικές μας συζητήσεις. Άλλος κανείς θέλει λόγο. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης. Της κυρίας Μαριέλ Γκάλο. Έχουμε την προστασία ε, ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους των τελωνιακών αρχών. Παρακαλούμε κυρία Γκάλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων του τελωνιακού κανονισμού κατά της παραποίησης και απομίμησης που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική, Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει φυσικά και το σχέδιο δράση των τελωνίων κατά της παραποίηση για την περίοδο 2009-2012. Θα ήθελα να σας επισημάνω μερικά αριθμητικά στοιχεία που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου τρέχοντος έτους που δείχνουν πραγματικά το εύρος ε, και τις διαστάσεις του προβλήματος. Ε, γίνεται αρκετή φασαρία στην αίθουσα, παραπονιέται η, η συγγήτρια. Ο αριθμός λοιπόν ε, των, κατασχέσεων που έκαναν τα τελωνία διπλασιάστηκε το 2010 σχέση με τα προηγούμενα χρόνια γιατί περ, περάσαμε από τα 43.500 στα 80.000. Μάλιστα οι κατασχέσεις ε, στα ταχυδρομικά δέματα πέρασαν από τις 15.000 το 2009 σε 43.000 και το 2010. Μάλιστα, η πρωταρχική κατηγορία κατασκευθέντων προϊόντων είναι σιγαρέτα 34%, ε, οικιακές συσκευέ 14,5% και στις οικιακές συσκευές στις ε, οικιακά προϊόντα που περιλαμβάνονται σαπούνια, παιχνίδια, αντικείμενα ένδυσης κτλ. 7%. Εδώ διακυβεύεται δηλαδή η υγεία και η προστασία των συμπολιτών μας. Στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να σας κάνω μία σύντομη επισκόπηση των ε, προτινόμενων τροποποίησεων του κανονισμού 1383 του 2003 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνω κάποια σχόλια για τις προτάσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή καταρχήν ε, του κανονισμού. Η διευρυμένη, η πρόταση παρατείνει το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού του 2003 και περιλαμβάνει τα εμπορικά ονόματα, τις τοπογραφίες των ημιαγωγών και τα, τους τρόπους χρήσης. Και συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής και κάποιες παράλληλες εισαγωγές, καθώς και κάποιες ε, συσκευές προκειμένου να παρακαμφθούν τα τεχνικά μέτρα. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό του 2003. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις παράλληλε εισαγωγέ, είχαμε ήδη μία ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Επιτροπή συγγνώμη, ΙΜΚΟ ε, εσωτερική αγορά για το θέμα αυτό και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Μια και στι ε, περισσότερε περιπτώσει η αυτούργοι αυτών των παράλληλων ε, εισαγωγών συμμετέχουν και στην απομίμηση παραποίηση προϊόντων. Για να αποφευθεί λοιπόν η υπερφόρτωση του έργου των τελωνιακών αρχών, θα πρέπει να διατίθεται η απαραίτητη τεκμηρίωση και πληροφορίες ώστε να μπορούν οι τελωνιακοί να εξακριβώνουν το κατά πόσο ένα προϊόν αποτέλεσε αντικείμενο παράνομης παράλληλης εισαγωγής. Σε ό,τι αφορά το, πεδίο εφαρμογή. ο αποκλεισμός των εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα που, που περιέχονται στις ε, προσωπικές αποσκευές, η εξαίρεση αυτή διατηρείται και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την εξαίρεση. Τέλος, ό,τι αφορά την, ε, το εμπόριο φαρμάκων και αυτή η διαμετακόμιση αποκλείστηκε από τον κανονισμό και αυτό για να αποφευχθεί μία αντιδικία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Βραζιλίας Ινδίας στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Σημειώνω αυτή τη συμφωνία, λαμβάνω υπόψη, αλλά γνωρίζοντας τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και γνωρίζοντας ότι τα ψευδοφάρμακα τα νοθευμένα φάρμακα κυκλοφορούν σε πολλές αφρικανικές χώρες και σε ασιατικές χώρες ή χώρες Λατινικής Αμερικής, δηλαδή σε χώρες που η οικονομία τους διέρχεται μια μεταβατική περίοδο, εκεί είναι που κυκλοφορούν τα περισσότερα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την πραγματικότητα και εμείς να τη λάβουμε απόψη. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο. Μετά το πεδίο εφαρμογή, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, το δεύτερο σημείο αφορά την απλουστευμένη διαδικασία καταστροφή αυτών των ε, προϊόντων. Πρόκειται για μια νέα πρόταση που καθιστά υποχρεωτική την απλουστευμένη διαδικασία καταστροφής των προϊόντων και προβλέπει κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ένα τεκμήριο συγκατάθεση, συνένεσης για τα παραποιημένα προϊόντα και προϊόντα πειρατείας, κάτι που επιταχύνει τη διαδικασία και την απαλλάσσει από γραφειοκρατικές διατυπώσεις, κάτι που θα μας ε, εξοικονομήσει πολύ χρόνο. Ένα τρίτο σημείο που καλό θα να συζητηθεί αφορά τα μικρά δέματα. Συμφωνώ απόλυτα με την αρχή της εισαγωγής ειδική διαδικασίας για τα μικρά δέματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους τρόπους εφαρμογής της, περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει όμως ε, να οριοθετήσουμε προσεκτικά αυτή την έννοια των μικρών δεμάτων, μικρών αποστολών. Και έχουμε και την παράγραφο 5 που χρήζει κάποιας εξέτασης γιατί προβλέπεται μια προθεσμία 20 ημερών για να συμφωνήσει ο δηλών ότι συμφωνεί με την καταστροφή του προϊόντος. Αν θέλουμε μία απλουστευμένη διαδικασία, τότε θα πρέπει να προβλέψουμε βραχύτερη προθεσμία. Η 20ήμερη προθεσμία είναι υπερβολικά μακροχρόνια. Επίσης, το θέμα της ευθύνης των τελωνιακών αρχών είναι ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Η υποχρέωσή τους ε, να δώσουν κάποιες εξηγήσεις σε περίπτωση καταστροφής. Και τελευταίο σημείο αφορά τις ε, δικονομικές εγγύσεις. Η νέα αυτή πρόταση προβλέπει κάποιες σημαντικές δικονομικές διαδικαστικές εγγύσεις, προβλέπει ε, τις διορίες παρακράτησης των ύποπτων προϊόντων, διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τελωνιακές αρχές θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον δικαιούχο τις πληροφορίες για τα δέματα, για τα προϊόντα και επίσης ε, μιλά για τις διαδικασίες που επιτρέπουν την καταστροφή των προϊόντων υπό τον έλεγχο των τελωνιακών αρχών σε περίπτωση ε, υποτιθέμενης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, το δικαίωμα υπεράσπισης ακρόασης ε, του κατηγορουμένου επίσης εξασφαλίζεται. Όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών θα πρέπει να γίνουν σεβαστά αλλά θα πρέπει να αποφευθούν χρονοβόρες και παραληπτικές διαδικασίες. Γιατί κάτι τέτοιο θα διακυβεύσει τον πρωταρχικό στόχο της πρότασης, της νομοθετικής αυτής πρότασης. Γιατί ο πρωταρχικός στόχος είναι η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των ε, επιχειρήσεών μας. Και επίσης η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Όπως ξέρετε, τρεις είναι οι ενδιαφερόμενες επιτροχές, οι επιτροπές, η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή, ο κ. Κρόιτσμαν είναι ο εισηγητής έκθεσης και οι επιτροπές ε, ΙΝΤΑ και Γιούρι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί ακόμη διαπραγματεύση μεταξύ των τριών επιτροπών. Η ΙΜΚΟ έχει προβλέψει χρονοδιάγραμμα να ψηφίσει την έκθεση Κρότσμαν στις 28 Φεβρουαρίου του 2012. Στη δική μας επιτροπή εγώ θα καταθέσω το σχέδιο γνωμοδότησής μου το Νοέμβριο ώστε να ψηφίσουμε στην πρώτη μας συνεδρίαση του 2012. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζω ότι δεν είναι και πολύ χλιδάτο αυτό το θέμα των τελωνίων. Ένας λόγος παραπάνω να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Γκαλό. Ο Σάσος Περώνης ζήτησε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την συνάδελφο για την ε, παρουσίαση της σύγησής της και να θέσω δύο ερωτήματα. Ένα, σχετικά με την ανάγκη ε, επιτάχυνσης των ε, πρακτικών καταστροφής των εμπορευμάτων, γιατί βεβαίως η ταχύτητα είναι επωφελής προς όλους. Ρωτώ λοιπόν, γιατί σε αυτή την περίπτωση ή θα πρέπει να γίνεται για προστασία των επιχειρήσεών μας ε, ε, γιατί από τη στιγμή που βρίσκονται ήδη ε, μπλοκαρισμένα στα τελωνία ε, όλα αυτά τα προϊόντα, το αν θα καταστραφούν σε πέντε μέρες ε, ή ένα χρόνο δεν νομίζω ότι αλλάζει ιδιαίτερα την κατάσταση για τις επιχειρήσεις μας, γιατί έτσι κι αλλιώς θα εστρεβλώνεται το ανταγωνισμός εάν έφταναν τα προϊόντα αυτά ε, στην αγορά. Επομένως, ναι, βεβαίως πρέπει να καταστραφούν τα εμπορεύματα αυτά, αλλά ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να καταστρέφονται πολύ γρήγορα ε, για να προστατεύονται οι επιχειρήσεις μας. Δεύτερον, το κόστος καταστροφής βαραίνει την χώρα στην οποία προσπαθούν γίνεται προσπάθεια να εισαχθούν τα προϊόντα αυτά ή ε, στον έμπορο ο οποίος παράνομα προσπαθεί να εισάγει τέτοια ε, προϊόντα απομίμησης. Ε, Λιχτενμπέργκερ. Εγώ ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Αφενός για το ερώτημα των παραλλήλων εισαγωγών ήδη έχουμε κρίνει για το στην ψηφοφορία iBred 2 και εδώ πρόκειται για το εάν επιβάλλουμε ένα αυστηρό καθεστώς στις παράλληλες εισαγωγές στραφόμαστε κατά του ίντερνετ γιατί καμία φίρμα στο ίντερνετ δεν μπορεί να λάβει όλη την ευθύνη για όλες τις εισαγωγές που κινούνται μέσω αυτής. Γι' αυτό το λόγο τότε είχαμε τότε ψηφίσει διαφορετικά. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι το θέμα και ήδη έχει υπάρξει μια ψηφοφορία. Επίσης, δεύτερο, η ανάληψη του κόστους της καταστροφής είναι ένα σημαντικό και κέριο θέμα. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνουν βέβαια και ο Ευχαριστώ, κύριο Σένστρομ. Ήδη είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γκαλό, την οποία ευχαριστώ, αλλά και δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια ζητήματα. Το πρόβλημα με αυτόν τον κανονισμό είναι ότι ξεπερνάει τον ουσιαστικό νόμο σε πολλά θέματα. Δίνει στα τελωνία ε, το δικαίωμα να κατάσχει νομίμως εισαχθέντα προϊόντα. Αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα και η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Δηλαδή, ε, το παράλληλη οι παράλληλε ε, είναι νόμιμη εμπορική διαδικασία και επομένω η δυνατότητα, ε, να η δυνατότητα που δίνεται στα τελωνία να σταματήσουν τη συναλλαγή αυτή σημαίνει ότι γίνεται εδώ υπέρβαση του ουσιαστικού νόμου. Ε, ε, δεν είναι δυνατόν επομένως απλώς να δοθεί ε, μια απλή επέκταση δυνατοτήτων στο τελωνίο. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικό τρόπο και με ειδική νομοθεσία. Οι μικρές αποστολές τώρα. Είναι γεγονός ότι συμφωνούμε όλοι ότι βεβαίως η απομίμηση, η παραποίηση προϊόντων είναι κάτι κακό. Και βεβαίως ε, είναι καλό που προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτό το κακό εμπόριο. Σε μερικές περιπτώσεις, όχι στις περισσότερες, προβλήματα ε, που αφορούν την υγεία, τη δημόσια υγεία κτλ. Αλλά κυρίως ε, δημιουργείται οικονομικό πρόβλημα για τις εταιρείε. Τώρα, Εάν ένας ε, ε, ιδιώτης καταναλωτής αγοράσει παπούτσια Nike ας πούμε, δηλαδή που έχουν το λογότυπο ε, Nike, σημαίνουν δύο περιστάσεις. Είτε είναι θύμα εγκληματικής ε, ενέργειας ε, γιατί δεν ξέρει ότι δεν είναι πραγματικό Nike ή ξέρει ότι δεν είναι πραγματικό αλλά παρόλα αυτά θέλει να το αγοράσει. Ε, σε μερικές χώρες μέλη, όχι σε όλες, είναι παράνομο να αγοράσει κανείς προϊόν παραποίησης ε, όμως είναι νόμιμο το να αγοράσει κανείς κάτι στο διαδίκτυο και για ε, λόγους ε, απολύτως και, για λόγους που δεν μπορεί να κατανοήσει ο αγοραστής δίνεται η δυνατότητα στα τελωνία να κατασχέσουν αυτό το προϊόν το οποίο έχει αγοράσει και επομένως δημιουργείται έτσι μεγαλύτερο πρόβλημα ενδεχομένως. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον ε, ε, αγοραστή ο οποίος αγοράζει μέσω διαδικτύου και τελικά φτάνουμε ε, στην αντίθετη όχθη. Ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Κανείς. Ενδεχομένως η εισηγήτρια θέλει να απαντήσει, θέλει να ολοκληρώσει την παρουσίασή της. Ε, ναι, κύριε Ανταλό, Θα ήθελα να πω δύο λόγια στον συνάδελφο Σπερώνη για να απαντήσω στα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που υπέβαλε. Βεβαίως ε, υπάρχουν ε, διαδικασίες αποζημίωσης των επιχειρήσεων Όσον αφορά το κόστος, όσον αφορά το κόστος καταστροφής είναι το άρθρο 27 που ασχολείται με το θέμα αυτό. Στην ουσία ε, αναλαμβάνει το κόστος αυτό ο υπόχρεος αλλά έχει δυνατότητα προσφυγής ε, κατά του εργοστασίου το οποίο παρήχθησαν τα παραποιημένα προϊόντα. Ε, συνήθως βέβαια τα προϊόντα προέρχονται από την Κίνα ή από άλλες ε, πολύ μακρινές και πολύ λίγο συνεργάσιμες ε, χώρες και επομένως εκεί έγκυται η μεγάλη δυσκολία. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των παραλλήλων εισαγωγών, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αξίζει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ε, είναι ένα ζήτημα λοιπόν επί το οποίο θα πρέπει να σκύψουμε με προσοχή. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για παράνομες, μιλάμε εδώ δηλαδή για τις παράνομες παράλληλες εισαγωγές. Μίλησα ήδη με, πολύ, με πολλούς ε, ε, ανθρώπους που μου είπαν ότι τις περισσότερες φορές οι παράνομες εισαγωγές ε, ε, βρίσκοντος στα ίδια φορτηγά και στα ίδια κοντέινερς με τις παράνομες ε, εισαγωγές, παράλληλες εισαγωγές, μαζί οι, παρά, οι παράλληλες εισαγωγές και νόμιμες και παράνομες. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θέλει να μιλήσει. Δεν φαίνεται να επιθυμεί κάτι τέτοιο. Επομένως, ολοκληρώσαμε και το σημείο 12 της κυρίας Μαριέλ Γκαλό. Και θα δώσουμε τώρα στον συνάδελφο λόγο στον Γιάνν Φιλίπ Άλμπρεχτ σχετικά με το δικαίωμα ε, σε ε, ε, δικαστική αρρωγή, σε δικηγόρο, όσον αφορά την ποινική διαδικασία δικαίωμα επικοινωνία μετά τη σύλληψη. Ευχαριστώ. Πρόκειται για πρόταση μέτρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της προσπάθειας να δημιουργηθούν κοινέ προδιαγραφές στο διαδικαστικό δίκαιο που έχει αρχίσει η προσπάθεια αυτή ήδη με τα θέματα μετάφρασης και διερμηνίας στην ποινική διαδικασία συνεχίστηκε με την οδηγία για το λεγόμενο Letter of Rights όπου υποτίθεται ότι εναρμονίζεται το δίκαιο περί των δικαιωμάτων και τώρα έρχεται το επόμενο μέτρο δηλαδή πρόσβαση σε δικηγόρο στην ποινική διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι όπως και ολόκληρο σε αυτός ο δικός χάρτης για το Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά σημαντικό μέτρο. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη έχουμε ζητήσει την εναρμόνιση και τη δημιουργία αυτών των κοινών προδιαγραφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Για παράδειγμα, όταν λήφθηκαν μέτρα αμοιβαίας αναγνώρισης σε ζητήματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, διακομματικά η αντίδραση ήταν θετική μέχρι τώρα και πιστεύω ότι πρόκειται για πρόταση που ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστεί να εκφράσουμε ως Νομική Επιτροπή την άποψή μας και να συμμετάσχουμε ως Κοινοβούλιο να δώσουμε εγκαίρως ως Νομική Επιτροπή τη γνωμοδότησή μας και να μπορέσει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών έτσι ώστε η διαδικασία να μπορέσουμε έγκαιρα να συνοδεύσουμε τη διαδικασία. Βρίσκω ότι είναι σημαντικό, διότι ήδη το Συμβούλιο Υπουργών έχει διεξαγάγει τις πρώτες συζητήσεις για την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Είναι λοιπόν σημαντικό το Κοινοβούλιο που συμμετέχει ομότιμα σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδικασία να μπορεί να προβαίνει σε σχολιασμό. από έξι χώρες μέλη του Συμβουλίου, μαθαίνω ότι αυτές είναι πολύ επιφυλακτικές απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν, μεταξύ άλλων, λόγω του ότι διότι οι δυνατότητες προστασίας του ατόμου πρόκειται να εναρμονιστούν σε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτήν ε, υιοθετεί το, το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ ορισμένες χώρες μέλη δεν συμμερίζονται την άποψη αυτή. Εγώ βρίσκω ότι η εναρμόνιση σε υψηλό επίπεδο είναι απαραίτητη και ως Ευρωβουλή θα πρέπει να πούμε καθαρά ότι επιθυμούμε τα δικαιώματα των ατόμων στην ποινική διαδικασία να εναρμονιστούν τουλάχιστον στο επίπεδο που αναγνωρίζει τα τελευταία χρόνια και με την ομολογία του έχει δημιουργήσει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται και ορισμένες παραπομπές που ζητούν παρόμοιες διατυπώσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε συνήγορο, όπως αυτές που έχει διατυπώσει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ιδίως τονίζω, βέβαια, τη δυνατότητα της προβολής και χρήσης αποδεικτικών στοιχείων. Τι από αυτά θα εξαρτάται, επίσης εάν έχει τηρηθεί η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συνήγορο Νομίζω ότι αυτά για το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι απαραβίαστα όρια, διότι όπως είπα ως Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε να μην υπάρχει πρόσβαση σε συνήγορο χωρίς να θεωρήσουμε ότι θα πάσχει η ανάκριση. Διότι αλλιώς τα πρόσωπα, εν προκειμένου οι ύποπτοι, δεν έχουν απολύτως καμία δυνατότητα αντίδρασης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να διατυπωθούν και αυτά τα για μας απαραβίαστα όρια. Έχω και την πρόταση για τις τροποποιήσεις που θα ζητήσει η Νομική Επιτροπή, για παράδειγμα για την θέση των παιδιών ή άλλων προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, Σε ορισμένα σημεία καθιστούμε σαφές ότι οι εξαιρέσεις λόγω εθνικών ιδιαιτεροτήτων γενικά από εμά δεν μπορούν να γίνουν δεκτές εφόσον τέτοιες ιδιαιτερότητες οδηγούν στην αποδυνάμωση των διατάξεων που πρόκειται να εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπου λοιπόν υπάρχει ασάφεια θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να εξαιρούνται οι ιδιαίτερες περιστάσεις των εθνικών δικαίων. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ένα επίπεδο εναρμόνισης, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν και ορισμένε αλλαγέ στα εθνικά δίκτυα. Σε ορισμένου τομεί. Βεβαίω, πολλέ χώρε ανταποκρίνονται ήδη σε πολλέ από τι προδιαγραφέ αυτέ, άλλωστε το καθιστά σαφέ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά, για μας είναι σημαντικό βέβαια να καταδείξουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε πολλές εξαιρέσεις στους κανόνες, αλλά να καθορίσουμε βασικούς κανόνες, βασικές αρχές που να μπορούν να εφαρμόζονται. Και οι εξαιρέσεις να παραμείνουν εξαιρέσεις. Έστω και αν σε ορισμένου τομεί αποδεικνύονται απαραίτητες. Και το λαμβάνουμε υπόψη αυτό στις τροπολογίες μας. Αλλά όπως είπα θα πρέπει οι εξαιρέσεις αυτές να περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο. Λοιπόν αυτές είναι ορισμένες από τις τροποποιήσεις που προτείνω. Βεβαίως με χαρά θα ακούσω ιδίω από τις σκιώδεις εισηγήτριες οι οποίες δυστυχώς είναι απούσες όλες σήμερα. Θα προσπαθήσω όμως την επόμενη εβδομάδα να οργανώσω μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών αλλά ελπίζω και από τους άλλους συναδέλφους της Νομικής Επιτροπής να λάβω σχετικές συμπληρώσεις, πολύ ευχαρίστως και τροπολογίες. Είμαι αρκετά ανοιχτό. Πρόκειται λοιπόν για μια πρώτη κατάθεση ιδεών, προτάσεων και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω κάνει και τις πρώτες επαφές με τους άλλους και και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε ταχαίως προς την κατεύθυνση σύνταξης μιας γνωμοδότησης και αναμένω βεβαίως τη συνεργασία σας. Ο κύριος Στογιάνοφ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω και τη γνώμη του εισηγητού βέβαια και να με διορθώσει αν ε, κάνω λάθος, αλλά εδώ ουσιαστικά μιλούμε για το δικαίωμα να κάνει ο κατηγορούμενος το γνωστό τηλεφώνημα, γιατί αυτό προβλέπουν συνήθω τα συντάγματα, ότι ο καθένας δικαιούται να κάνει τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να συνεχίσετε. Στις ε, αμερικανικές ταινίες, στον αμερικανικό κινηματογράφο, βλέπουμε αυτό το δικαίωμα να κάνει κανείς το τηλέφωνο. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συζητούμε εδώ σήμερα. Και ας με διορθώσει ο εισηγητής, αν κάνω λάθος. Το βουλγαρικό σύνταγμα προβλέπει ότι ο συλληφθής έχει δικαίωμα σε πρόσβαση σε δικηγόρο και μάλιστα από τη στιγμή της σύλληψής του. Βέβαια, αυτά προβλέπει το Σύνταγμα, η θεωρία. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Πριν από μία τριετία συνελήφθη και χωρίς να ληφθεί υπόψη η βουλευτική μου ασυλία, με συνέλαβαν, μου έβαλαν χειροπέδες, με κλώτσαν στο κεφάλι, στην πλάτη. Πώς να υπερασπίσει κανείς τα δικαιώματά του με τέτοια μεταχείριση. Παρόλο που επαναλαμβάνω τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται σε πολλά έγγραφα ότι ο κάθε κατηγορούμενος, ο κάθε συλληφθής έχει δικαίωμα ε, πρόσβαση σε δικηγόρο, δικαιούται να κάνει τα τηλεφωνήματα κτλ. Η πράξη είναι τελείως διαφορετική. Στις αμερικανικές ταινίες βλέπουμε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να κάνει ένα τηλεφώνημα. Όταν εγώ συνελήφθη, δεν είχα καν δικαίωμα Δεν ε, μου απαγγείλθηκε καν κατηγορία. Όλα μου τα δικαιώματα παραβιάστηκαν. Όλα αυτά λοιπόν τα δικαιώματα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στα διάφορα έγγραφα που εγκρίνουμε. Και δεν θα πρέπει μόνο να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα, αλλά να περιλαμβάνονται και σχετικές προθεσμίες. Όταν με συνέλαβε η βουλγαρική αστυνομία, η διορία ήταν 24 ώρη. Δεν ξέρω θεσμία και στις άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν τα δικαιώματα του συλληφθέντος να αναφέρονται ρητά στα έγγραφα που, που καταρτίζουμε. Και τι δικαίωμα Επικοινωνία έχει επίσης συλληφθεί, με ποιου. και όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τον κύριο Άλμπρεχτ στη σύνταξη τη έκθεσή του και στην επιτυχία της έκθεση αυτής, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία, όπω σα είπα, με σύλληψη, παρόλο που δεν είμαι και ιδιαίτερα περήφανο γι' αυτή. Ο Σέλφο Περόνι. Ευχαριστώ. Βρήκα όμως το έγγραφο την απάντηση στην ερώτηση που ήθελα να υποβάλω, οπότε άλλες ερωτήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννα Άλμπρεχτ, τον εισηγητή για την έκθεσή του, καθώς επίσης και για τα καλά λόγια, για τους επένους που απίθυνε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επαφής ε, με ε, ε, τρίτο άτομο σε περίπτωση σύλληψης είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό η ουσιαστική πρόσβαση σε δικηγόρο τελικά ε, δίνει νομιμότητα σε όλη την ε, ποινική διαδικασία και διασφαλίζει την δίκαια δίκη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρατε ήδη, προβλέπει το, την δυνατότητα κάθε ε, κρατούμενου να έρθει σε επαφή με τρίτο πρόσωπο, διπλωματική αποστολή κτλ. Ε, για οποιονδήποτε έχει ε, συλληφθεί είτε είναι πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι. Έχουμε επίσης ε, και την ε, απόφαση Φάλντος 2008 του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδεικνύει σαφώς, αναφέρει ρητά ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης θα πρέπει να, τα πάντα να γίνονται παρουσία δικηγόρων. Επίσης ε, αποσαφηνίζονται τα πάντα ξεπερνώντας ενίοτε και την ε, ε, νομολογία του δικαστηρίου άρθρα 5 και 6 πρόκειται για άρθρα τα οποία δεν προβλέπονται από την νομολογία του δικαστηρίου. Επίσης όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει παρουσία του δικηγόρου ε, και για τις ε, διαδικασίες ε, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Αυτό βεβαίως ξεπερνάει και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως η πρόταση ξεπερνάει και την ομολογία και κατά κάποιο άλλο στοιχείο. Δηλαδή περιγράφει ας πούμε τις δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να ασκήσει εξ ονόματος του πελάτου του ο δικηγόρος. Ε, σύμφωνα με την πρότασή μα λοιπόν ο δικηγόρο πρέπει και μπορεί να παίξει ενεργητικό ρόλο, ε, να είναι παρόν σε οποιαδήποτε ανάκριση, να θέτει ερωτήσεις και να ζητά αποσαφηνήσει. Θα πρέπει ε, να είναι επίσης παρόν στην, σε περίπτωση μαρτυριών ή σε περίπτωση συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Η πρόταση προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα ε, στα, στις ανάγκες της έρευνας και στα δικαιώματα της υπεράσπισης. Και μονάχα σε εξαιρετικέ περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε ε, δικηγόρο. Μονάχα δηλαδή σε περίπτωση που με τον τρόπο αυτό ε, προστατεύεται καλύτερη η ανθρώπινη ζωή. Η πρόταση προβλέπει και μία σημαντική διάταξη ε, όσον αφορά στις αποζημιώσεις ε, σχετικά με παραβίαση ε, της, του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο. Δηλαδή, ε, τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσπαστεί χωρίς την παρουσία δικηγόρου και ε, με ε, παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο, αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ, δεν είχα να πω τίποτα άλλο για την ώρα και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Πρόεδρος, ολοκληρώσαμε την εξέταση. Α, όχι, ο κύριος Άλμπρεχτ. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ο κύριος Άλμπρεχτ, ο εισηγητής. Ναι. Δεν θέλω να επιμικίνω ανώφελα τη συζήτηση, όμως ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αντιδράσω σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαρθρωθούν η θεωρία και η πράξη στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις χώρες μέλη είναι ότι υπάρχουν κάποιες αρχές ε, οι οποίες ε, ορίζονται ε, από τις συνθήκες, από την νομοθεσία κτλ. Αλλά η πρακτική δεν είναι πάντα καλή. Εκεί έχουμε και καλά πρότυπα, καλά παραδείγματα, αλλά και λιγότερο καλά. Επίσης ε, έχουν υπάρξει μέτρα όπως ας πούμε η εμιβαία αναγνώριση, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, που προσπαθούν να εναρμονίσουν κάποιες καταστάσεις. Αλλά κατά την άποψή μου θα είναι αναπόφευκτο ε, να ε, δημιουργηθεί ως ονούπο ένα ελάχιστο ε, όριο το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλες τις χώρες. Ξέρουμε βεβαίως ότι μετά άλλες χώρες μπορούν να, να μεγαλώσουν αυτό το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και ε, ε, εκεί θα πρέπει να δούμε εάν ε, το, κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με τέτοιες διαδικασίες διαφοροποιημένες ή εάν ε, θέλουμε να έχουμε ε, ε, πραγματικά εξίσωση προς τα κάτω γιατί ξέρουμε ότι συχνά οι αστυνομίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να δουν ποιες είναι οι χείριστες πρακτικές και όχι οι βέλτιστες. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εξίσωση προς τα κάτω. Ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται παντού και επίσης να σιγουρευτούμε ότι ε, είτε μιλάμε για την Βουλγαρία είτε μιλάμε για την ε, Γερμανία είτε για οτιδήποτε θα πρέπει να γίνονται σεβαστές αυτές οι διαδικασίες, οι ποινικέ, ε, τις οποίες, οι οποίες διασφαλίζονται δια νόμου. Και επίσης ένα δεύτερο στοιχείο, επιχείρημα, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι το εξής Εάν σε μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπέγραφε την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τότε, τότε είναι πιθανό ε, η προκείμενη περίπτωση να αποτελεί δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στρασβούργου ε, και επομένως ε, τελικά να βρει ας πούμε αντίκτυπο στα συντάγματα των χωρών ή ε, αν θέλετε ε, στα, στα δικαϊκά συστήματα των χωρών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλεγεί για να εφαρμόζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους ε, την εφαρμογή τους λέγω από τις χώρες μέλη. Ο κύριος Στογιάννοφ ξαναζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποιους ελάχιστους κανόνες, ελάχιστες προδιαγραφές και παρέμβαση του δικηγόρου κατά την πρώτη ανάκριση του υπόπτου. Πάντως, περισσότερες χώρες μέλη το habeas corpus δεν εφαρμόζεται. Ενώ σε κάποιες χώρες εφαρμόζεται το habeas corpus. Και μάλιστα πριν ε, την πρώτη ανάκριση. Ερωτώ λοιπόν, δεν θα έπρεπε ο δικηγόρος να είναι παρόν από την αρχή ή ακόμη και πριν από την πρώτη ανάκριση. Πριν ε, απαγγελθεί κατηγορία δηλαδή, ώστε να μπορεί να βοηθήσει ο δικηγόρο στην ε, εφαρμογή του χαμπέας κόρπους. <clears throat> Ωραία, ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε επ' αυτού. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 14. Η συγγήτρια είναι η κυρία Εύα Λίχτενμπέργκερ. Όμω, Όμω δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, διότι εσείς προτείνετε, ε, προτείνετε ψηφοφορία, γιατί η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 5 και επομένως δεν μπορούμε ε, να ξεκινήσουμε πριν από τις 5 την ψηφοφορία. Μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας και μετά όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε. Uh, I was... uh, Ich um, kann ja Deutsch reden. Entschuldigung. <laughs> Καλύτερα να μιλήσω γερμανικά. Probleme. Um, die... Κύριε Πρόεδρε, έχουμε το θέμα της πρόσβασης στα διάφορα έγγραφα πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, φυσικά η βασική αρχή εδώ που θα πρέπει να πριτανεύσει κατά την εξέταση της πρότασης είναι η αρχή της διαφάνειας. Προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση αλλά τώρα η Επιτροπή προτείνει ένα ταχύτερο ρυθμό από αυτό που αρχικά είχαμε προβλέψει. als, ε, hintergrund, ε, sehen, dass das schon... Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία της ανάκτησης παλιάς πρότασης. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια νέα πρόταση με ένα πολύ μικρό τμήμα της αρχικής. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτή την συρρυκνωμένη πρόταση, γιατί θεωρούμε ότι χρειάζεται μια γενικότερη πρόταση που φοβόμαστε ότι δεν θα ευοδοθεί. Ο κύριος Κάσμαν προτείνει την συνοπτική διαδικασία. Επίσης ε, σκεφτήκαμε να ε, επιταχύνουμε τη διαδικασία στέλνοντας μια επιστολή. Φαντάζομαι ότι αντίγραφο της επιστολής ε, έχετε λάβει όλοι. Αλλά στο μεταξύ άλλαξαν οι προθεσμίες και παρόλα αυτά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δεχτείτε αυτή την επιστολή γιατί πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα την επιδίνωσε το blackout που είχαμε την περασμένη φορά και δεν μπορέσαμε να συνεδριάσουμε. Χάσαμε και από εκεί χρόνο. Βέβαια το blackout ήταν ουσιαστικά περίπτωση ανωτέρας βίας, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο αν δεχτούμε την επιστολή. Θέλει κανείς το λόγο? Όχι. Επομένως, σας προτείνω να σταματήσουμε για 15 λεπτά και να ξαναρχίσουμε στις 5 παρα 5. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξαναρχίσουμε. Θα ψηφίσουμε πρώτα Μάλλον όχι, να το θέσω διαφορετικά. Συζητήσαμε το σημείο 14 με την ε, εισήγηση που μας έκανε η κυρία Εύα Λίχτενμπέργκερ και από τη στιγμή που πέρασε η 17η απογευματινή μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση της ε, Εύα Λίχτεμπερκ, πρόσβαση, ε, δημόσια πρόσβαση στα ε, έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ. Chi vota Κατά. Astenuto. Αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνεται πάντως. Περνάμε τώρα στο επόμενο. Ψηφοφορία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Η συγγήτρια η κυρία Νταϊάννα ε, Βόλις, την οποία θερμά καλωσορίζουμε γιατί ξέρετε πόσο μακρινά, μακριά από την Ευρώπη είναι η Αγγλία και γι' αυτό ε, άργησε να έρθει. Αστειεύομαι βεβαίως. Ναι, ναι και παρόλα αυτά ε, φυσικά σας καλωσορίζω θερμότατα. Προχωρούμε λοιπόν. Εναλλακτική επίλυση διαφορών. Alternative Dispute Resolution. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υμκο Β. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. εγκρίνεται ΙΜΚΟ-ΔΙ Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. εγκρίνεται ή Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ίμκο F, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά. Ε, όχι, μισό λεπτό. Ε, ε, ανεβοκατεβάσατε υπερβολικά γρήγορα τα χέρια σας. Ψηφίζουμε την τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 7, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 7, τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, υπέρ. Κατά. να μετρήσουμε. Ε, παρακαλώ πολύ να ξαναψηφίσουμε. Δεν έγινε καλά η καταμέτρηση. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. ΥΜΚΟ 7. Δεύτερο τμήμα όχι δεν θα το ψηφίσουμε. Πάμε στο, στην τροπολογία ΙΜΚΟ 18, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 2, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 8, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 10 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ίμκο 11 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ίμκο 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ίμκο 20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. να ξαναψηφίσουμε. Ήμκο ε, 20. Υπέρ. Ήμκο 20. Εγκρίνεται. Αλλά πριν έγινε λίγο διαφορετική η ψηφοφορία. Κατά εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για την υπόδειξη. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ήμκο 3 πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο υπέρ κατά αποχές ομόφωνα κρίθη η έκθεση. Περνάμε τώρα στην έκθεση Λένε σχετικά με τη Σύμβαση των Αθηνών. Μεταφορά, θαλάσσια μεταφορά επιβατών και ε, αποσκευών. Ε, μία ψηφοφορία μόνο. Υπέρ, κατά, αποχές. Ομόφωνα είναι κρίθηκε αυτό. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Μέντερς είναι γνωμοδότηση σχετικά με τον αθλητισμό. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Καρύμ υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία Μάντερς υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 <coughs> υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 και συμβιβασμός ταυτόχρονα μάντερς υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος υπέρ κατά 2-3 καταψηφίζετε ναι. Τέλερ, Νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβουμε την ε, ψηφοφορία γιατί η Φρανσουάς δίστασε λίγο και μας μπέρδεψε. Ψηφίζουμε λοιπόν ο, επί του συνόλου της γνωμοδότησης υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. και μία αποχή. Και μία αποχή από τον κύριο Σπερώνη. Λοιπόν, θα σταματήσουμε για τρία λεπτάκια, γιατί μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. C'è Lopez Royo. Dispute involving Parliament. Questo è a porte chiuse. Ah. Porte chiuse. Se, se le può dire che il resto lo votiamo. Il resto lo votiamo a porte chiuse. Comincia la riunione a porte chiuse.